Λοιπόν, ε, Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο πρόεδρος έλαβε έτοιμα να οριστεί η κυρία Πιτέρα στη θέση της κοινίας Κοσλόφσκα στην αντιπροσωπεία σχέσεων με τη Λευκορωσία και στην κοινοβουλευτική συνέλευση.